Okay, everybody, we'll open the meeting and start it. Άρχεται η συνεδρίαση. Αν τα πάμε γρήγορα μπορούμε να κάνουμε και ένα διάλειμμα πριν από τις ε, ψηφοφορίες. Οπότε, πρώτα απ' όλα μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Θέλετε κάποια αλλαγή, όχι. Οπότε περνάμε στις ανακοινώσεις της ε, Προέδρου σημαντικό αυτό γιατί ενημερώνω την κατάμεστη επιτροπή για το τι έγινε στον τριμερή διάλογο. Από την τελευταία μας συνεδρίαση είχαμε πολλές ε, τριμερείς διαλόγους για εθνικούς και περιφερειακούς λογαριασμούς. Μετά υπήρχε και την δεύτερη συνάντηση. Πολλές καλές συμβιβαστικές λύσεις στο διατακτικό μέρος. Το παράρτημα Α έχει σχεδόν κλείσει. Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί 21 ή 22 Ιουνίου και αφορά το παράρτημα Β, οδηγία Omnibus 2. Εκεί πέρα είχαμε κάποια πρόοδο, είχαμε άλλη μια συνάντηση αρχές αυτής της εβδομάδας, αλλά ο βασικός στόχος, δηλαδή η ευθυγράμμιση της φερεγγιότητας 2 με τον ΑΙΟΠΑ 2 δεν επετεύχθη. Η Κομισιόν έχει μια πάρα πολύ περιοριστική άποψη όσον αφορά τις προδιαγραφές παρά το ότι αυτό έχει γίνει ήδη σε άλλες οδηγίες. Η Κομισιόν λοιπόν έχει προσκληθεί στις 20 Ιουλίου στην επόμενη συνάντηση. Έχουμε επίσης ένα εκτιμώντας για το δημόσιο χρέος, την ανάγκη για πίνακες συσχετισμού και το ζήτημα των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και εγγυήσεων. Επίσης, αυτή την εβδομάδα είχαμε τον πρώτο τριμερή διάλογο για Ευρωπαϊκά Ταμεία Επιχειρηματικού Κινδύνου και Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αυτοί οι διάλογοι γίνονται από κοινού επειδή άλλοι επικαλύπτονται τα δύο θέματα πρώτη ανταλλαγή απόψεων έγινε για τις τροπολογίες Συμβουλίου και της δικής μας Επιτροπής και η επόμενη συνάντηση προγραμματίζεται 12 Ιουνίου στο Στρασβούργο. Επίσης, αυτή την εβδομάδα είχαμε δύο τριμερείς διαλόγους για την Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 4 και το CRR. Ακόμα Βεβαίω είμαστε στην οδηγία και σε θέματα σύνταξης για επίμαχα ζητήματα και προσπαθούμε να επιτύχουμε συμφωνία για τα λιγότερο επίμαχα. Θα συνεχιστεί λοιπόν η δουλειά, πολλές ακόμα τριμερείς συναντήσεις ε, μεταξύ των οποίων και σήμερα το απόγευμα και στο Στρασβούργο την άλλη εβδομάδα. Αυτά λοιπόν για τους τριμερείς διαλόγους. Νομίζω πως ε, αυτή τη στιγμή στις ανακοινώσεις θα ήθελα να αναφέρω πως ε, μου είπες ε, την προσοχή στο ότι έχουμε κάποια περίεργα email από πλευράς λόμπι που συμπεριλαμβάνουν μέχρι και βίντεο. Σβέν, για πες μας. Ναι, ήθελα να πω πως θεωρώ πως η αποστολή ε, βίντεο σκριν ε, που στέλνουν ένα μήνυμα ε, παραπάει δηλαδή είναι βίντεο και ήχος που δεν μπορεί κανείς να, να σταματήσει εντάξει μου τα στέλνουν χάρτινα και τα ρίχνω στην ανακύκλωση δεν ξέρω αν το έλαβαν και άλλοι συνάδελφοι καλό ήταν να περιοριστεί ο κόσμος ε, στα χάρτινα και στα απλά ηλεκτρονικά μηνύματα και όχι στα ηλεκτρονικά σκουπίδια. Έλεος δηλαδή. Το να μας στέλνουν ηλεκτρονικά πράγματα χωρίς να μας ρωτάνε δεν βοηθάει ούτε την ουσία ούτε το περιβάλλον. Μάλιστα. Θα έχουμε ψήφισμα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, λοιπόν. Περνάμε στο σημείο 3. Ανταλλαγή απόψεων για μήνυ οδηγία για την ευθυγράμμιση των ημερομηνιών για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας ε, στην οδηγία Omnibus 2 χωρίς ε, να έχουμε κάποιο νομοθετικό κενό για ζητήματα ασφαλιών. Εγώ είμαι η συγγήτρια. Ε, εξορισμού γιατί γίνεται με απλοποιημένη διαδικασία για να μην έχουμε λοιπόν νομικό κενό όταν θα ε, δημοσιευτεί μετά τις 31 Οκτωβρίου 2012 η οδηγία αυτή η Κομισιόν προτείνει η ημερομηνία εφαρμογής ε, της ε, οδηγίας φερικιότητας στις 36 του του 13 και την ημερομηνία επιβολής στον ε, έκτο του 14. Αυτά τα συμφωνήσαμε στον τριμερή διάλογο, αλλά για να μην βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου θα έχει σταματήσει να ισχύει η φυστάμενη οδηγία και δεν θα έχουμε νέα οδηγία ενισχύ, πρέπει να αλλάξουν οι οδηγίες. Οπότε θα έχουμε μια οδηγία με τρεις γραμμές μόνο, τρεις σειρές, για να γίνει ακριβώς αυτό. Συμφωνήσαμε με τους συντονιστές και τη διαπραγματευτική ομάδα της Omnibus 2 να το εγκρίνουμε χωρίς τροπολογίες. Αλλά βεβαίως είμαι υποχρεωμένη να ενημερώσω την Επιτροπή στην περίπτωση που κάποιος θέλει να σχολιάσει. Ο Μπέρκχαρτ, ο εισηγητής για το θέμα δεν είναι εδώ, αλλά έχουμε ήδη συζητήσει στον τριμερή διάλογο πως θέλουμε να ε, γίνει αυτό. Θέλει κάποιος να σχολιάσει, όχι, ωραία, μπράβο θα κάνουμε αυτό το οποίο σας είπα για να μην έχουμε νομικό κενό. Σημείο 4. Το σημείο 4 αναβάλλεται. Το 4 θα ήταν το πρώτο θέμα για τους οργανισμούς αξιολόγησης ε, και τώρα περιμένουμε να έρθουν οι υπόλοιποι. Οπότε κάνουμε ένα μικρό interlúdio, γύρω στα 10 λεπτά διάλειμμα.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 Έχετε τις κάρτες, έχετε βάλει να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Right, happy buttons to be pressed. We've only got 28. Λοιπόν, μόνο 28 μέλη παρόντα έχουμε, μόνο. Oh, we've got 32 now. That's getting better. 33. 32-33 βελτιωνόμαστε. Right, come on, press your buttons to make sure it works. We've got 34 cards plugged in and 29 Έχουμε 34 κάρτες που είναι μέσα στη... Αλλά δεν έχουν πατηθεί όλα τα κουμπιά. 35 κάρτες έχουν πατήσει το κουμπί 31 άτομα τέσσερις κάρτες μέσα στη θέση τους, αλλά δεν έχουν πατηθεί τα κουμπιά τα ανάλογα. Σάρων αν είναι έλκυ είναι εντάξει, ακούγεται από κάτω. Σας το λέω αυτό σε περίπτωση που κάποιος πατάει ένα κομβίον, θεωρεί ότι λειτουργεί, αλλά δεν λειτουργεί. Και αυτό είναι σημαντικό, ότι δουλεύει το κουμπί. There are still three, three... Ε, τρεις κάρτες στη θέση τους, αλλά τα κουμπιά τα αντίστοιχα δεν έχουν πατηθεί. Yeah, but I wonder where it is, though. I mean, it... okay. There's only one. There's... Right, 36. 36 λοιπόν κάρτες με 36 κουμπιά πατημένα. Το ξέρω ότι άμα σας πρόξω θα το κάνετε. 32 είναι ικανοποιημένοι, 4 δεν γνωρίζουν. Είμαστε έτοιμοι να κινήσουμε λοιπόν. Άντολιν Σάντσες Πρεσέδο η έκθεσή του για την υπόθηκα δάνεια είσαστε όλοι έτοιμοι Αντολίν πρέπει να ξεκινήσουμε Ξεκινάμε την έκθεσή σου Αντολίν Πρώτα απ' όλα ο τίτλος ΙΜΚΟ 1 υπέρ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 στη σελίδα 9 του αγγλικού συμβαστική D λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική αλφα ε, ΑΚ στη σελίδα 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική G1 στην επόμενη σελίδα είναι όλες συμβαστικές τροπολογίες λέει προφορικές τροπολογίες στο κείμενό σας επειδή υπάρχουν πολλές ομάδες ε, λέει συμβαστική αλλά δεν αλλάζει το κείμενο Λοιπόν, τι κάνω. Ξεκινάω από τη συμβαστική G πρώτα και μετά συμβαστική G2 που είναι η προστίκη. Συμβαστική G πρώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το συμπληρωματικό κομμάτι το G2 υπέρ το κομμάτι που ήταν προφορική τροπολογία τώρα αποκαλείται συμβαστική G2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στη συμβαστική H στη σελίδα 17 Όλα τα ροζ είναι συναρμοδιότητες και περνάνε αυτόματα. Συμβιβαστική H λοιπόν. Πρώτα απ' όλα έχουμε προφορική τροπολογία. Λοιπόν, του ECR υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική H υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική γιώτα στη σελίδα 21. Ξεπερνάμε όλα τα ροζ κομμάτια που ήταν τη ΣΥΜΚΟ. Και εδώ οι προφορικές τροπολογίες έχουν μετατραπεί σε τμήματα. Ποιο τμήμα ήταν το έκτο. Η, η προφορική τροπολογία γίνεται το έκτο τμήμα της συμβαστικής. Αλλά το κείμενο είναι το ίδιο. Αυτή τη σειρά θα ακολουθήσουμε έξι τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται. Καλύτερα να κάνουμε έναν έλεγχο σε αυτό το δεύτερο τμήμα. απορρίπτεται 17 υπέρ 21 ψήφι κατά τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίθηκε αλλά ας γίνει έλεγχος για την ε, μικρή διαφορά ψηφίσατε όλοι ευχαριστώ εγκρίνεται 21-17 Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Αν, μπορείτε να, αν μπορούσατε να ψηφίσετε στις ίδιες, με την ίδια προσέγγιση, ίδιες ομάδες. Ψηφίσατε όλοι. Άλλος ένας να ψηφίσει. Εντάξει, πέρας. Απορρίπτεται. 17 υπέρ, 20 ψήφοι κατά. Πέμπτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έκτο τμήμα που ήταν προφορική τροπολόγια υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά θα κάνουμε έναν έλεγχο για το έκτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ, 22 ψήφοι κατά. Ερμήνευα διαφορετικά τη ψηφοφορία μιας ομάδας πριν. Πάμε στην τροπολογία 492, στη σελίδα 30. ...492 λοιπόν υπέρ... ...κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική K στη σελίδα 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική L στην επόμενη σελίδα αποτελείται από τρία τμήματα Πρώτο τμήμα λοιπόν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη βαστική μη στη σελίδα 37 το αγγλικού κειμένου σε τέσσερα τμήματα. Συμβαστική M λοιπόν, μη, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Μπορούμε να ελέγξουμε αν θέλετε το δεύτερο τμήμα. Έλεγχος λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 22 κατά, οπότε απορρίπτεται τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος και εδώ. Τρίτο τμήμα, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτεται. 18 με 20. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική νη στη σελίδα 43 του αγγλικού κειμένου φτάσατε εκεί πρώτα απ' όλα έχουμε προφορική τροπολογία και μετά τρία τμήματα αυτή τη σειρά θα ακολουθήσω πρώτα απ' όλα λοιπόν την προφορική τροπολογία να προσθεθούν από τη διαδικασία διάθεσης πιστώσεων υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Είναι αρκετά μικρή διαφορά. Ψηφίσατε όλοι πέρα ψηφοφορίας, απορρίπτεται 16 υπέρ με 21 ψήφους κατά, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ας γίνει ένας έλεγχος για το τρίτο τμήμα που νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται πραγματικά. 18-20. Συμβαστική όμικρον στη σελίδα 45. Όχι, λάθος. Στην προηγούμενη σελίδα είναι. Έχουν προφορική τροπολογία που αντικαθιστά την τελευταία φράση υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Συμβιβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική π στη σελίδα 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q στη σελίδα 46 τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο τμήμα θα ήταν να ελέγξουμε τι έγινε στο δεύτερο τμήμα λοιπόν ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα Τρία τμήματα έχουμε εδώ. Θέλω να σας διαβάσω. Μόνο δύο τμήματα ακούγεται, έτσι δεν είναι. Όχι, τρία τμήματα λέει η Πρόεδρος. Να σας διαβάσω λοιπόν. Πρώτο τμήμα, το κάναμε αυτό. Δεύτερο τμήμα, τα κράτη-μέλη μπορούν να απαγορεύσουν τη χρήση του όρου συμβουλή, συμβούλου, ανεξάρτητη συμβουλή κλπ. κλπ. Και λέει να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο τέλος. Τρίτο τμήμα μετά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιτρέψουν μόνο τη χρήση του όρου ανεξάρτητη συμβουλή ή ανεξάρτητο σύμβουλο όταν οι διάφοροι ε, πιστωτές κλπ. κλπ ε, που, εκεί που λέει που αμείβονται δεν αμείβονται κλπ. Το έχετε αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το τρίτο τμήμα ε, στον κατάλογο ψηφοφορία. Α, είναι, το, είναι πρωινός κατάλογος, είναι πρόσφατος. Με το πρωινό ήρθε δηλαδή η πρόεδρος. Α, είναι στη βραδινή εκδοχή. Ο εισηγητής μας θα πρέπει να μας πει πώς θα ψηφίσουμε. Είναι σημαντικό. Ψηφίζουμε πρώτο το δεύτερο τμήμα. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Θα κάνουμε τον έλεγχο, λέει ο πρόεδρος. Δεν θέλετε να δείτε ποιο είναι το δεύτερο και το τρίτο τμήμα. Έχετε το κείμενο. Το έχετε. Να τσεκάρετε, να δείτε τι λένε τέλος πάντων. Το δεύτερο τμήμα θα ήθελα. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Λοιπόν, πρώτο τμήμα, καλά τα πήγαμε. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα, λέει η Πρόεδρος τώρα. Ψηφίσατε όλοι το δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας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 κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R3 στην επόμενη σελίδα. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική, όχι, τροπολογία 135 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική S σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική ΤΑΦ στη σελίδα 55 πρώτα μια προφορική τροπολογία του ΕΛΚ που την υποστηρίζει άλτε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δύο τμήματα έχουμε για το υπόλοιπο. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική W στη σελίδα 57 ξεκινώντας με την προφορική τροπολογία που την υποστηρίζει το L και το ΑΛΤΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έχουμε μετά το συνολικό κείμενο. Συμβιβαστική W στο σύνολό της υπέρ. Δεν είναι κατά τμήματα, δεν είναι κατά τμήματα. Αναφέρονται την παράγραφοι, αλλά δεν είναι κατά τμήματα. Δεν είναι προφορική τροπολογία. Λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική, στην επόμενη σελίδα, όχι Συμβιβαστική διπλό α, αλφα α, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 156 στην επόμενη σελίδα. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα αν θέλετε. Μου φάνηκε ότι τα κάθε το απορρίφθηκε. Τέλο πάντων. Λοιπόν, δεύτερο τμήμα τη συμβαστική ΑΑ, έλεγχο. Λοιπόν, ψηφίσατε. Τέλος ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται 14 με 22. Νομίζω πως εδώ πέρα μπροστά παραδιασκεδάζεται. Λοιπόν, στην 156 είμαστε υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. 156. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 20 υπέρ 16 κατά. Συμβαστική ΑΒ με προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά εποχές. Απορρίπτει προφορική τροπολογία. Συμβαστική ΑΒ όπως ήταν υπέρ κατά εποχές. Δεκτή. Συμβαστική AC στην επόμενη σελίδα. Υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική AD Είναι με, η 726 είναι με άσπρο. Ο κατάλογος μου είναι λάθος. Μάλιστα. Ψηφίζουμε την τροπολογία 726 και τις υπόλοιπες. Υπέρ κατά αποχές δεκτές 164 100, 160 καταπίπτει μάλιστα ΙΜΚΟ 112 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ανδρέας νομίζω ότι είσαι υπέρ ε. Συμβαστική AD υπέρ κατά αποχές Δεκτή. Περνάμε τώρα στην 165. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι είναι δεκτή. Να επαληθεύσουμε την 165. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ, 19 κατά. Ήμκο 114, ε, πρώτη παράγραφος υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 7.30 και γιούρι 53 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 7.31 και οι παρομοίες υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Εφτά υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι είναι δεκτή αλλά να την επαληθεύσουμε 7.36 και 115 ΙΜΚΟ Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ 20 κατά. Οπότε περνάμε τώρα στην 737 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται περνάμε στη συμβαστική αε στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές δεκτή ΙΜΚΟ 122 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να το επαληθεύσουμε ΙΜΚΟ 122 στο κάτω μέρος σελίδας 63 Α, μια στιγμή. Α, καταπίπτει. Μάλιστα, οπότε έχει καταπέσει. Ε, την απορρίψαμε ούτως ή άλλως, οπότε τα ίδιο κάνει. Και περνάμε στην 764. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 765 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. Θα έλεγα ότι είναι 7.65 επαληθεύουμε. Καταπίπτει με ισοψηφία. Ήμκο 123 υπέρ. Κατά αποχές. Εκτή. 866 υπέρ κατά αποχές δεκτή ίδια με ΙΜΚΟ και Γιουρί συμβαστική AF σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε τώρα συμβαστική C σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε τώρα στην 768 σελίδα 70 μου ξέφυγε κάτι στο μισό. Συμβαστική μη. Okay. Right. This is... Μάλιστα. Ε, είναι από αυτά τα περίπλοκα. Δηλαδή, εάν εγκρινόταν η συμβαστική C μαζί με την RHQ, M και N, περνάμε στην συμβαστική 768 και όχι στην R γιατί η R θα ψηφιστεί μόνο εάν δεν γίνει δεκτή κάποια από όλες τις άλλες. Οπότε περνάμε στην 768 σελίδα 70. They did all carry, yeah, presumably. They did, I checked. I've got a list Mr. Gozes has a point. Yeah, Jean-Paul. Jean-Paul. Je, n'ai pas fait l'école, je n'ai pas... Εγώ δεν έχω βγάλει το Πολυτεχνείο, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω. Στην 66 εσείς έχετε διαφορετικές σελίδες. Συμβιβασμός H λέει συμβιβασμός H θα εγκριθεί εάν ο συμβιβασμός H έχει εγκριθεί. Κοιτάξτε, από τότε που πήρε η αριστερά την εξουσία στη Γαλλία δεν καταλαβαίνουμε πια τίποτα. Να, το εξηγήσω, να το εξηγήσω. Άμα το εξηγήσετε κιόλας, θαύμα. Μα πρέπει, πρέπει κανείς να είναι υπηκό βασιλείου για να το, Υπηκό βασιλείου για να το εξηγήσει Τι εννοεί. Η συμβαστική AIDS περιέχει διατακτικό και εκτιμώντας. Αυτά είναι τα εκτιμώντας του AIDS. Και αντί να μην είναι στον κατάλογο της ψηφοφορίας, είναι στη σειρά τους μεταξύ των εκτιμώντων, αλλά στην πραγματικότητα έχουν καλυφθεί με την συμβιβαστική. Γιατί έχει γίνει δεκτή η AIDS. Κοιτάξτε, πρέπει να το λύσουμε, γιατί αλλιώς ο κόσμος θα αρχίσει να αναρωτιέται τι εστί Ευρώπη. Εγώ θέλω να εξηγήσω ότι αυτό το τρίτο άρθρο του συμβιβασμού σε είναι ορισμοί και τους ορισμούς τους έχουμε εγκρίνει στις άλλες τρεις δράσεις. Γι' αυτό λοιπόν τη συμπεριλαμβάνουμε εδώ. Είναι αναφορά των προηγουμένων δράσεων. Η μέθοδος που ακολουθήσαμε είναι να θέσουμε τους ορισμούς στο πλάι για να μπορούν όλοι να παρακολουθούν γιατί αυτά τα τρία ζητήματα θα μπουν στις ε, πράξεις συνδιαλλαγής. Όλα καλά, όλα καλά. Προσπαθήσαμε απλά να έχουμε κάποια διαφάνεια. Και τώρα προσπαθούμε να ψηφίσουμε την 768. 768. Υπέρ. Περιμένετε. Στη σελίδα 70 ήταν, Ζαν Πολ. 768 υπέρ κατά αποχές δεκτό 126 της ΣΥΜΚΟ υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική AG υπέρ κατά αποχές δεκτή τώρα περνάμε στην AA που είναι ακριβώς από κάτω Against. κατά αποχές δεκτή AH στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική α στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε τώρα στη συμβαστική β έχουμε εδώ πέρα μια νέα χωριστή ψηφοφορία, να το διαβάσω αν δεν το έχετε. Το πρώτο μέρος είναι το εκτιμώντας 8 τελευταία περίοδος που λέει άρα αυτή η οδηγία θα πρέπει να ισχύσει για την εγγύηση πίστοση στους καταναλωτές αλλά τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την ε, ισχύ σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που δεν είναι καταναλωτέ δηλαδή μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με την ε, οδηγία 263 του 2003 για τις ε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος είναι το υπόλοιπο. Το βρήκατε. Μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μέρος δεύτερο το υπόλοιπο εκτιμώντας το 8, 9, 10 και 10α υπέρ κατά αποχές δεκτό συμβαστική C στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές δεκτό περνάμε στην επόμενη AJ υπέρ AI Α, είναι σκοτεινό και δεν το διαβάζω. AI υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τώρα περνάμε στην AJ υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Μετά περνάμε στην συμβιβαστική IHN και W. Μάλιστα. Συμβαστική συμβιβαστικών. Αυτά μου αρέσουν υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. Συμβιβαστική AB υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μετά περνάμε στην ΑΚ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μετά πάμε σε άλλη μία στις EFGS, τις συμβιβαστικές. Τι είναι? Μάλιστα. Από ό,τι μου λένε, εγκρίνονται αυτές αυτομάτως. Πρόκειται για αυτόματη ε, συμβιβαστική τροπολογία που εγκρίνεται από μόνη της. Νομίζω πως οι σκιώδεις ηγητές έχουν να ξέρουν τι συμβαίνει. Ναι, είναι πολύ, είναι πολύ εύκολο. Ξέρετε πως στην οδηγία ε, κεφαλιακών απαιτήσεων 3 ήμασταν κατά των ε, πολύ πολύπλοκων ε, προϊόντων αλλά τώρα απορρίφθηκαν αυτά και έχουμε τώρα το πακετάρισμα του πακεταρίσματος τώρα θα τα βλέπουμε στην επόμενη αναθεώρηση της οδηγίας την 5 ή την έκτη μάλιστα πρόκειται για τίτλοποιημένη δηλαδή τροπολογία αλλά έχει εγκριθεί ωραία ο Αντελίν μάλλον ξέρει πως είναι σωστό. Περνάμε τώρα στην I, στην επόμενη σελίδα, υπέρ, κατά αποχές δεκτή, συμβαστική K, η οποία εγκρίνεται αυτομάτως, επειδή είχε εγκριθεί η K. Μα, γιατί είναι το, το εκτιμώντας που πήγαινε με το προηγούμενο. Οπότε εντάξει, δεκτή. Okay, the, come on, let's, let's... Μάλιστα. Λοιπόν, α, ε, ας, ας σοβαρευτούμε. Συμβαστική L, L. Υπέρ. Χωριστή ψηφοφορία. Είστε σίγουροι, <laughs> κυρία Πρόεδρε. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ναι, ναι. Α, ε. άμα χαχανίζει και η πρόεδρος δεν τα πάμε καλά. Λοιπόν, τώρα έχουμε άλλο ένα εκτιμώντας που εγκρίνεται από μόνο του και περνάμε συμβαστική όμικρον. Ναι. Ναι, ναι, Κυρία Πρόεδρε, έχω την εντύπωση ότι άμα πραγματικά κινηματογραφείται αυτή η συνεδρίαση θα έχει μεγάλη επιτυχία στα μαργαριτάρια που προβάλλει τηλεόραση στο τέλος της χρονιάς. Κοιτάξτε, έτσι και τα ανεβάστε στο YouTube έχουμε βρει τον πελά μας. Και δεν βλέπω τώρα κιόλα. Λοιπόν, συμβαστική O που ε, εγκρίθηκε από μόνη της, οπότε περνάμε στη συμβαστική N εκτιμώντας, τα οποία από και αυτά από μόνα τους εγκρίθηκαν. Ε, η κυρία Πρόεδρε εδώ πέρα μοιάζει με τις αυτόματες συναλλαγές. Και η N είναι αυτόματη, γιατί πρόκειται για τα εκτιμώντας της ίδιας, το αυτό και για την P. Ε, λοιπόν, για να ψηφίσουμε, η επόμενη είναι... Συγγνώμη. Υπάρχουν δύο M για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση. Έχουμε δύο συμβαστικές M. Okay. hang on. Can we, can we just clarify compromise M? ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει πρόβλημα με την M υπήρχαν δύο συμβαστικές μη Εγώ ήθελα να εξηγήσω ότι όταν εγκρίναμε τα, μεμονωμένα άρθρα παρουσίαζα ταυτόχρονα και το εκτιμώντας και το άρθρο. Γι' αυτό είχαμε λοιπόν κάθε φορά δύο τμήματα. Επειδή εγκρίναμε εμείς τους, τους συμβιβασμούς πριν από τα άρθρα, με το Recite πήγαινε ο συμβιβασμός. Γι' αυτό τώρα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι δεδομένα. Διότι όλοι οι εγκεκριμένοι συμβιβασμοί έχουν τα αντίστοιχα άρθρα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα συνάφειας. Όποιος συμβιβασμός πέρασε, πέρασε. Γιατί ο κάθε συμβιβασμός έχει Και έχετε εκτιμώντα δίπλα. Μάλιστα. Μέχρι το AF θα πάμε τώρα στο κάτω της σελίδα 83. Όλα αυτά μέχρι εκεί είναι εκτιμώντα που αντιστοιχούν στα άρθρα τους και έχουν υιοθετηθεί μαζί με τα αντίστοιχα άρθρα. Για να μην λοιπόν έχουμε άλλο γέλιο πάμε στο τέλος της σελίδας 83 και τη σημαστική AF υπέρ λοιπόν κατά αποχές δεκτό και τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε το κείμενο ολόκληρο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε ψήφισαν όλοι ωραία πέρας 35 υπέρ 3 κατά μια αποχή ηλεκτρονική πλειοψηφία ηλεκτρονική με ψηφοφορία επί του νομοθετικού ψηφίσματος ψήφισαν όλοι πέρας 35 υπέρ 2 κατά 2 αποχές Yes, yes, Sven. Oh, I think. Okay. Um, I'm told we have got a very Λοιπόν, έχουμε ένα κατάλογο πολύ πιο ήρεμο και ήμερο το σχέδιο γνωμοδότησης του Τίοντορ Στόγιον για την εφαρμογή της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη. Ε, είστε όλοι έτοιμοι. Ξεκινάμε. Συμβαστική α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές. Ένεχος για την 7. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται 16 με 22. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 τροπολογία 6 μάλλον συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται No, that was rejected. So we need to do the original. Can we? 18. I think. Sorry, 18. Yeah, 17 was the same. Η 17 ήταν ταυτόσημη. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο κατά πίπτη. Λοιπόν, τροπολογία 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές έλεγχος λοιπόν επαλήθευση για την 22 Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 20 με 17. Τροπολογία 23 που είναι προφορική τροπολογία. Προφορική τροπολογία τροπολογίας. Προφορική τροπολογία πρώτα που αφορά την τροπολογία 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και τροπολογία τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία του τροποποιημένου κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. 38 υπέρ. Καμία ψήφος εναντίον. Καμία αποχή. Πολύ καλά τα κατάφερε Οπότε τελειώσαμε. Η επόμενη συνεδρίαση είναι τη Δευτέρα 11 Ιουνίου